everybody. Καλώς ήρθατε. Ας αρχίσουμε με αυτό το τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Το πρώτο σημείο που έχουμε είναι γνωμοδότησή μας στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Η ΑΦΕΤ με τον Πέτρα Αστρεβίτσιους, είναι επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή και ο δικός μας συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Φάρια που έφτασε, οπότε μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το σημείο. Οι σκιώδη ηγητές δεν βλέπω να είναι εδώ, θα είναι σύντομη συζήτηση, τι να κάνουμε, αλλά το βασικό είναι να σα ακούσουμε για να μας εισάγετε κάπως το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, ήταν τιμή μου που ανέλαβα τη σύνταξη γνωμοδότηση όσον αφορά την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Η έκθεση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο είναι κάτι που ενδιαφέρει και την Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέρφους. Ακόμα δεν έχουμε συναντηθεί με τους σκιώδεις εισηγητές γιατί είμαστε στην αρχή της διαδικασίας. Σίγουρα όμως θα ακούσω πολλές προτάσεις από τους σκιώδεις εισηγητές, τους συναδέρφους μας. Προς το παρόν, ευχαριστώ πάντως για τη στήριξή σας που μου αναθέσατε τη σύνταξη της γνωμοδότησης αυτής. Από... Θα ευχαριστήσω την κυρία Ρίτα από τη Γραμματεία της Επιτροπή μας και την κυρία Βερζινέκλιν από το ΕΛΚ Σύμβουλο για την βοήθειά τους. Χωρίς αυτή τη βοήθεια θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για μένα. Μόλις έφτασα σε αυτήν την επιτροπή, δεν ήμουν πριν μέλος, οπότε καταλαβαίνετε ότι η βοήθεια αυτή είναι πολύτιμη. Έχουμε λοιπόν διάφορες προτάσεις που ζητάμε να συμπεριλάβει η ΑΦΕΤΕ στη δικιά της έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017. Το σχέδιο αυτογνωμοδότησης πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, κυρίως με τους στόχους 3 και 5, όπως επίσης και με την Ατζέντα 2030 πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία Spotlight, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΟΗΕ, ώστε να καταργηθεί κάθε μορφή βία σε βάρος των γυναικών. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι όπως γνωρίζουμε, οι Ηνωμένε πολιτείες φαίνεται να παρεκκλίνουν από τις παγκόσμιες στρατηγικές, οπότε και από αυτές τις δύο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πάντως στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας, είναι από τους κύριους παράγοντες στήριξης. Δεν μας στηρίζουν όλες οι χώρες του ΟΙΕ, αλλά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτιέρες, ναι, και είπε ότι η επένδυση στις γυναίκες είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπος για την ε, ανύψωση των ε, κοινωνιών. Το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης χωρίζεται σε τρία κομμάτια, θα έλεγα. Το ένα είναι η καταπολέμηση της βίας και η πρόληψή της. Το δεύτερο είναι η καταπολέμηση των καταναγκαστικών γάμων και το τρίτο είναι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην ε, εκπαίδευση. Από ό,τι φαίνεται, πολλές γυναίκες ήταν θύματα σεξουαλικής βίας από πολύ νωρίς, άρα πρέπει να φροντίσουμε ακόμα περισσότερο για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Επίσης πρέπει να υπάρξει περισσότερο συνδυτοποίηση για την καταπολέμηση της ενδοικογενειακής βίας, που εξακολουθεί και παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι χώρες μέλη θα πρέπει επίσης να κυρώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πολλές χώρες έχουν ήδη κυρώσει τη σύμβαση αυτή, όχι όμως όλες. Για να καταπολεμηθεί ακριβώς αυτό το φαινόμενο γιατί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και η απάλληψη των διακρίσεων είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες κακές πρακτικές πρέπει να εξαφανιστούν από παντού στον κόσμο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε παραδείγματα που αναφέρονται στις παραδόσεις, στις θρησκευτικέ ή άλλες. Οι συστάσεις του ΟΗΕ είναι ξεκάθαρες. Τα κορίτσια έχουν το δικαίωμα στην παιδική ηλικία και πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τη ζωή τους όπως επιθυμούν. Η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης πρέπει να φροντίσει για αυτές τις αρχές. Μέσα από όλες τις ε, δράσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το κάνει αυτό και στις διαπραγματεύσει που έχει με τρίτες χώρες. Αγαπητοί συνάδελφοι, γι' αυτό Σα είπα ποιε είναι οι προτεραιότητε, καταπολέμηση τη βία, καταπολέμηση των κανακαστικών γάμων και πρόθεση τη εξίσου πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτά τα τρία στοιχεία ζητάω να συμπεριλάβει αφέτη στην έκθεσή τη. Επιπλέον, τονίζω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα στον κόσμο. Ίσως εσείς να διαβάσατε ήδη το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Έχω συμπεριλάβει λοιπόν δύο περιπτώσεις δύο εξτρεμισμού που είναι για τους Θωρίκα και για τη Βενεζουέλα. Η Ροχίνκα και η Βενεζουέλα. Αυτές είναι δύο περιπτώσεις όπου έχουμε μια πολύ διακατάσταση στον κόσμο. Πρόκειται για ανθρωπιστικές τραγωδίες σε βάρος των κοινοτήτων αυτών, αλλά μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο αν δεν γίνει τίποτα. Συνεπώς, όσον αφορά την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις δύο αυτές περιπτώσεις, τους πρόσφυγες δηλαδή από τη Βενεζουέλα και την μειονότητα των Ροχίνγκια. Ξέρετε ότι οι δύο αυτές κοινότητες είναι ιδιαίτερα ευάλωτε στη βία κατά των γυναικών. Τα στοιχεία που έχουμε για αυτές τις δύο κοινότητες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Γι' αυτό η εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτέ τις περιπτώσεις. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σα τι απειλές αυτές σε βάρο των γυναικών και μάλιστα όχι μόνο για τώρα αλλά ακριβώς επειδή ξέρουμε τι έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, γι' αυτό και η σύσταση αυτή πιστεύω αποκτά μεγαλύτερη ακόμα σημασία. Περιμένω λοιπόν τις παρατηρήσεις τα σχόλια των συναδέρφων και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας για να προχωρήσει αυτός ο σημαντικός φάκελος και να συμπεριληφθούν οι προτάσεις μας στην έκθεση της ΑΦΕΤ. Όντως είμαστε στο πρώτο στάδιο. Θα υπάρξει χρόνος για προτάσεις από τους συναδέρφους και από τους κοιόδης ηγητές. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει έρθει η ώρα να λάβουν το λόγο σκιώδεις εισηγητές. Η ε, κυρία Ward έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή εδώ. Ε, ήμουν στα εγγένεια της πλατείας Κόξ. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή για τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων και εκπροσώπησα το Κοινοβούλιο. Η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών θεωρεί πως η γνωμοδότηση είναι αρκετά καλή, απευθύνεται και αντιμετωπίζει τα περισσότερα ζητήματα ισότητας, και θα υποβάλουμε ορισμένες τροπολογίες έτσι ώστε να δώσουμε έμφαση στις σεξουαλικές μειονότητες και τα δικαιώματα των ε, ΛΟΑΤΚΙ και άλλα θέματα. Όπως γνωρίζετε το Συμβούλιο εξεδόσε κατευθυντήριες γραμμές ε, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις κατά τον ΛΟΑΤΚΙ και η ομάδα S&D θεωρεί πως είναι πολύ σημαντικό αυτές οι κατευθυντήρε γραμμές να εφαρμόζονται και η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να δείχνει ευαισθησία ως προ τα δικαιώματά του. Θέλουμε ιδιαίτερα να ασχοληθούμε με την κατάσταση ε, που βιώνουν οι χείρε ε, στι περιοχέ που πλήττονται από ένοπλε συγκρούσει και επί τη ευκαιρία να πω ότι θα συμμετάσχω σε ένα συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον κοινωνικό αποκλεισμό ε, και τις διακρίσεις που υφίστανται χείρες. Προσεχώς. Επίσης, ε, στις τροπολογίες θα προτείνουμε την προσθήκη κάποιων παραγράφων που δείχνουν πόσο σημαντική είναι και η πνευματική υγεία στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, θα θέλαμε μια εντονότερη διατύπωση των ε, σε των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και τέλος θεωρούμε ότι ο κοινωνικός ε, διάλογος ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, θα συνεισφέρει πολύ στην εξωτερική πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Να προσθέσω και να πω κιόλα πως εκτιμώ πάρα πολύ την ε, γνωμοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν θα ήταν δυνατόν να υπογραμμίσουμε το ρόλο των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία. διότι συνδέεται και αυτό με την ε, δημοκρατία, με την ειρηνευτική διαδικασία κτλ και είναι εξάλλου ένα θέμα που αν ε, μπορούσατε να το συμπεριλάβετε στη γνωμοδότηση, νομίζω πως θα την εμπλούτιζε. Θα δώσω τώρα το λόγο ξανά στον εισηγητή, αν θέλει να σχολιάσει. Ωραία, θα ξεκινήσω από το τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι άντως πολύ σημαντικό ε, να γίνει αναφερό σε αυτό, γι' αυτό θα περιμένω και τις προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να κυνηγήσουμε το όραμα αυτό. Ε, να σας πω βέβαια ότι το σκέφτηκα αυτό που είπατε. Και να σας πω επίσης ότι συναντήθηκα με ε, άτομα ε, εκπρόσωπους των Πεσμέργα και ε, με εξέπληξε αυτό που άκουσα είναι φανταστικό ε, αυτό που συμβαίνει, πολύ καλό το έργο τους και επίσης γνωρίζετε πώς είμαι προασπιστής των ε, δικαιωμάτων μειονοτήτων και ΛΟΑΤΚΙ. Ανήκω σε αυτήν την ομάδα ε, εργασίας. Να σας επιστήσω την προσοχή λοιπόν στο ότι αυτό είναι ένα προσχέδιο. Δεν είναι πλήρες ακόμα. Ελπίζω να το ολοκληρώσουμε τις ερχόμενες εβδομάδες. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα σεξουαλικά δικαιώματα, τα παραγωγικά δικαιώματα επίσης ε, είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών και τους ε, στόχους τους, μιλάμε για ισότητα των φίλων και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό εξάλλου είναι και ένα λεπτό ζήτημα, πολύ ευαίσθητο για πολλούς. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χωρίς ε, να ε, πατήσουμε κάλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ε, διαπολιτισμικό διάλογο, φυσικά και είναι σημαντικός και εκείνος, μπορώ να σας πω ότι Αυτό είναι και το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου εξάλλου, ο διαπολιτισμικός διάλογος και το λέω χωρίς να θέλω να ακουστώ έτσι υπερβολικά θρήσκος. Σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις σας και ε, προσβλέπω στην ε, καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Οπότε, πέραμε στο επόμενο σημείο ή όχι. όχι. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. 2 Οκτωβρίου έως τις 5 το απόγευμα. Ψηφοφορία στη ΦΑΜ. 22 Οκτωβρίου και στην ΑΦΕΤ 5 Νοεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για τροπολογίες και ψηφοφορίες. Οπότε, παίρνουμε τώρα πράγματα στο επόμενο σημείο προφορική ερώτηση σχετικά με την οπισθοδρομική αντίδραση στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φίλων. Κ. Λόπες, πολύ σημαντικό θέμα. Ήδη στη μικρή ομάδα είχαμε μια πολύ έντονη συζήτηση, οπότε ξεκινώ δίνοντα τον λόγο στον κύριο Λόπες, τον συντάκτη. Κυρία Πρόεδρε, θα ξυπήσω τους διερμηνείς για να μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα. Ας δούμε τα δύο κείμενα που συζητούμε σήμερα. Ε, ξεκινώ με μια εισαγωγική παρατήρηση. Το ψήφισμα που έχετε μπροστά σας ως κείμενο είναι τελές γιατί είναι, δεν είναι παρά ένα αρχικό κείμενο. Υπάρχουν και περιορισμοί όσον αφορά το μέγεθος του κειμένου με τους οποίους έπρεπε να συμμορφωθώ. Όμως, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την προφορική ερώτηση. Είναι μια καλή αρχή, πιστεύω, για να αναπτύξουμε το θέμα κατά τη διάρκεια της ζήτησης και να δούμε τι θα κάνουμε εν του ψηφίσματος στο οποίο τη συμβολή όλων περιμένω. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη, παρατηρούμε μια πιστοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Ατομικά, δικαιώματα στην υγεία, σεξουαλικά, αναπαραγωγή, εργασιακά κλπ. Παρατηρούμε μια υποχώρηση λόγω της υποβάθμισης του μέτρης της υγείας, της μείωσης της χρηματοδότησης εν γέννη. Το ίδιο βλέπουμε όσον αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, χειρότερη πρόσβαση σε αποβολές. Όλα τα δικαιώματα εν γέννη, λοιπόν, βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Γονεϊκά δικαιώματα κλπ. Η επίκληση της νομοθεσίας γίνεται όλο και πιο δύσκολα. Υπάρχουν δυσκολίες ε, όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα νεπιαγωγεία κλπ. Και στην εκπαίδευση, λοιπόν, και γενικότερα δεν υπάρχει σεξουαλική εκπαίδευση, ο κόσμος δεν διδάσκεται πώς να χρησιμοποιεί αντισυλληπτικά, προφυλακτικά και ούτω Εμείς αποβλέπουμε σε μια κοινωνία ισότιμου σεβασμού. Όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση, την καταπολέμηση θα έλεγα όλων των μορφών βία κατά των γυναικών. Τα πρόσφατα λοιπόν χρόνια τι παρατηρούμε. Παρατηρείται έξαρση αυτών των φαινομένων βία. ιδιαίτερω κατά γυναικών στην ηλικία τη εφηβεία. Πολλέ φορέ έχουμε βία στο σπίτι, παρενοχλήσει παρενοχλήσεις στο χώρο εργασία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δηλαδή πρέπει να αναζητήσουμε και τις αιτίε και να μελετήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις της βίας στο χώρο εργασία. Έχουμε μια περίπτωση στην Πορτογαλία, η οποία βγήκε στη δημοσιότητα πρόσφατα. Νομίζω είναι ένα το παράδειγμα, αυτό που λέω. εργατρία απολύθηκε παράνομα. Παρά το γεγονό ότι το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επανέλθει στην εργασία της. Επί μήνες όμως, τώρα, υποχρεώνεται να φορτώνει και να ξεφορτώνει την ίδια παλέτα με τα ίδια ακριβώς εμπορεύματα ε, στον ήλιο, στεκόμενοι εκεί επί ώρες. Ε, καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια άλλη μορφή βίας. Δεν είναι παρενόχληση, είναι βία ψυχολογική και σωματική βία κατά αυτής της ε, γυναίκας. Γι' αυτό για άλλη μια φορά λέω ότι πρέπει να κυρώσουμε αλλά και να εφαρμόσουμε ακόμη περισσότερο τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και δεν είναι ο μόνος μηχανισμός, το μόνο, μόνη η συμφωνία, το μόνο κείμενο που πρέπει να αξιοποιήσουμε σε αυτόν τον αγώνα στον αγώνα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών. Δυστυχώς γίνεται συστηματική προσπάθεια να αποκρυβούν αυτές οι διαφορές, αυτές, αυτά τα κρούσματα βίας. Πολλές γυναίκες ε, υποχρεώνονται εμέσως ή αμέσως να επιστρέψουν στο οικιακό περιβάλλον. Υφίστανται τις συνέπειες της ανεργίας. Ε, δυσκολεύονται να ξαναπροσεγγίσουν την αγορά εργασίας στο ψήφισμα υπάρχουν τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία που δεν καλύπτουν φυσικά τα πάντα. Θα προσθέσουμε και άλλα στοιχεία και περιμένω και τις δικές σας συνεισφορές. Είτε γραπτός, είτε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είτε με τη μορφή τροπολογιών. Επίσης, θέλουμε να αναφερθούμε στην επίπτωση της λιτότητας. Λιτότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για την ικανοποίηση αυτών των δικαιωμάτων στην πράξη. Υπάρχουν στη θεωρία, αλλά όχι στην πράξη. Εν κατακλείδη, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και του συνεργάτε μου. Συγγνώμη, μερικά ε, ονόματα δεν τα προφέρω καλά. Σας ευχαριστώ πραγματικά για όλη τη βοήθεια και για τα δύο κείμενα. Από εκεί πέρα είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Περιμένω και τις ε, τροπολογίες, έτσι πως θα προκύψουν από τη συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό ψήφισμα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Σκιώδης πρώτα και μετά οι άλλοι βουλευτές. ΕΛΚ, Αναμαρία Κουράτσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ανέτα. Εκ μέρους του Σκιώδους, του, της κυρίας Πυρκάινεν, ε, ζητώ συγγνώμη, κολλείεται όμως. Θα κάνω την μπορώ για να την ε, εκπροσωπήσω απαξίως. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ άνδρων και γυναικών. Δεν πρόκειται λοιπόν για επικουρικό ζήτημα, περιφερειακό ζήτημα. Η πρόοδος στον τομέα δεν είναι βεβαίως γραμμική. Οι σχετικέ προσπάθειες δεν πρέπει να χαλαρώσουν. Γίνονται αντιθέτω προσπάθειες ακύρωση αυτής της πρόοδου παγκοσμίω, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιστρομική αντίδραση είναι πολλές φορές ε, σημάδι κοινωνικών διαφορών. Απειλούνται όμω εν γέννη δημοκρατία και το κρατούς δικαίου. Συνεπώ, οποιαδήποτε τέτοια αντιδραστική κίνηση χρειάζεται να παρακολουθείτε στενά. Χρειάζεται ακόμη περισσότερο δράση, χρειάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση της. Κάποια νέα κρατημέλη, υπενθυμίζω, δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κατά της οικικής βίας, της βίας. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να υιοθετήσουν, να στερνιστούν ως προτεραιότητα τον στόχο της ισότητας. Τα, τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται από το Σύνταγμα, γιατί αυτό έχει σχέση με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Επίσης, τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία και μάλιστα κατά προτεραιότητα. Τέλο, πέρα από έναν χάρτη πορεία για την επίτευξη των στόχων μα μεταξύ αυτών την εξάλληψη κάθε είδου βία κατά των γυναικών. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά από τη Σκιωδή Συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Από τους σοσιαλιστές. Worth. Word. Παρακαλώ. Εγώ μιλώ εκ μέρου του Εντουάρ Μαρτά, ο οποίο δυστυχώ κολλείται για οικογενικούς λόγους, έπρεπε να επιστρέψει στη Γαλλία. Ζητά συγγνώμη. Θα διαβάσω το κείμενό του. Ευχαριστώ τον εισηγητή για δύο εξαιρετικέ προτάσεις, δηλαδή το ψήφισμα και την προφορική ερώτηση. Επιτρέψτε μου προς το παρόν να τονίσω δύο-τρία ζητήματα και θα τα συζητήσω με τον εισηγητή και τους κοιόδες στο μέλλον. Πρώτον, ερωτώ την Κομισιόν γνωρίζουν αυτήν την οπισθοδρομική αντίδραση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών. Τι κάνει η Κομισιόν. Λυπούμε, διότι απουσιάζει οργανωμένη αντίδραση κατά όλων των επιθέσεων κατά των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. Εν ώψη των προτάσεων του ΣΥΙΤΗ, ζητώ νομοθετικές προτάσεις με αυτό το αντικείμενο και δει για την αντιμετώπιση των ψευδοειδήσεων. Χρειάζεται ένα κεφάλαιο, ειδικά για τις ψευδοειδήσεις που αφορούν τις ε, αμβλώσεις και την αντισύλληψη. Σήμερα πολλοί Ευρωπαίοι αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες. Μάλιστα ένας ε, τέτοιο ε, νόμος κατά των ψευδοειδήσεων ψηφίστηκε στην Γαλλία πέρσι και έχει αποδώσει τα μέγιστα Συνεχίζει ο Ντουάρ. Μιλώντα λοιπόν για δικαιώματα και ισότητα, προτείνω μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για τα θύματα τη πορνεία, τα οποία θα τα βοηθήσει να ξεφύγουν από τον κλειό αυτών. Υπάρχουν διάφορε λύσει. Ε, Ένα κοινό τόπο θα ήταν να υποστηρίξουμε τα θύματα της πορνείας, επαναλαμβάνω, με ενισχύσεις, ε, με κονδύλια με εκμάθηση ξενών γλωσσών, ε, παροχή στέγη κλπ. Χρειάζεται λοιπόν ειδικό προπολογισμό. Ξέρω όμω ότι είναι πρόβλημα αυτό γιατί τα κρατημέλη βλέπουν τον προπολογισμό εν γέννη να μειώνεται. Αυτέ είναι οι γενικέ ιδέε του Εντουάρ, ε, τι οποίε θα χαρεί πολύ να συζητήσει μαζί σα. Ζητά συγγνώμη και πάλι Εντουάρ που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα μαζί μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Τζούλη. Δεν έχεις και εσύ το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ με απασχολεί εμένα και με ανησυχεί αυτό το έγγραφο που είναι προπαγάνδα και παρουσιάζει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση σαν να είναι η μοναδική σωστή. Όταν μιλάμε για τα ίσα δικαιώματα, παρακαλώ να σέβεστε και τις δικές μου απόψεις σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Εκτός αν θέλετε να έχετε μαζί σας μόνο τους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις με εσά. Αλλά δεν είναι αυτό δημοκρατία. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το έγγραφο αυτό προωθεί μια εικόνα της κοινωνίας σαν να είναι η μόνη σωστή. Μιλάμε εδώ πέρα για αυτή την οπισθοδρόμηση που είναι φεμινιστική ορολογία και που έτσι φαίνεται να είναι και ολόκληρο το έγγραφο. Έχει μια επικριτική και αρνητική εικόνα οποιοδήποτε έχει διαφορετική άποψη. Το έγγραφο δεν αφήνει περιθώρια για συζήτηση, ούτε για μια ευρύτερη παρουσίαση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες. αντιαποκρίνονται στους στόχους της αριστεράς τόσο αναφέρονται σε αυτό το κείμενο. Ε, ίσα δικαιώματα δεν σημαίνει ίδια ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να έχουν τα ίδια. Σημαίνει ότι η γυναίκα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ανθίζει σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους και πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Ακούστε με παρακαλώ. Είναι κρίμα που η άποψη που έχουμε εδώ παραβλέπει τα πραγματικά προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. Ας δούμε το θέμα της ε, γονικής άδειας, ε, της απελευθέρωσης στο, στη Γαλλία ή στο Βέλγιο. Είναι 15 με 16 εβδομάδες, αλλού είναι λιγότερο λιγότερο και από τέσσερι εβδομάδε. Στην Πορτογαλία, γιατί αναφέρατε την Πορτογαλία, είναι μόνο δέκα εβδομάδε. Μία γυναίκα η οποία στο τέλος της εγκυμοσύνης της δεν έχει καλή υγεία, δεν μπορεί να φύγει με αναρωτική έξι μήνες πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται ότι θα αρχίσει η μητρική άδεια. Οπότε έχει μόνο δύο μήνες στη διάθεσή της για να είναι με το παιδί της μετά τη γέννα. Άρα απομακρύνεται από το μωρό της ακριβώς τη στιγμή που εκείνο τη χρειάζεται περισσότερο, αλλά επιπλέον αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες που δεν είναι πολύ καλά στην υγεία τους αναγκάζονται να επιστρέψουν στην εργασία τους λίγο μετά τη γέννα. Κάτι το οποίο μπορεί να έχει συνέπειε στην υγεία της και την ε, σωματική και την ψυχολογική. Θα σας δώσω εγώ και κάποια παραδείγματα, αλλά δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν. Η περισσότερες γυναίκες υπάλληλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξέρετε ότι όταν ε, εγκυμονούν μπορούν να δουλέψουν γιατρικούς λόγους ε, με μερική απασχόληση. Αυτό όμω δεν είναι αρκετά γνωστό, γιατί η πληροφορία αυτή δεν κυκλοφορεί στους υπαλλήλου. Υπάρχει ένας άντρα στην αίθουσα αυτή που η γυναίκα του υπάλληλο εδώ έκανε τέσσερα παιδιά και δεν ήξερε ότι είχε αυτό το δικαίωμα. Γιατί ένα τέτοιο δικαίωμα, μια τέτοια πληροφορία δεν ε, διαδίδεται, αλλά αντίθετα κρύβεται. Αυτό είναι ο πιστοδρόμηση. Όταν δεν ε, αφήνουμε την γυναίκα να ενημερωθεί για τα δικαιώματά της, ότι μπορεί να δουλεύει δηλαδή πολύ λιγότερο από 8 ώρες δεν το γνωρίζουν οι γυναίκες και δεν το χρησιμοποιούν αυτό το δικαίωμα. Στην δήλωση διαβάζουμε για το δικαίωμα στην άμβλωση και ότι οποιο δεν συμφωνεί με αυτό δεν είναι προδευτικός. Όχι, δεν είναι προδευτική αυτή που περιορίζονται στα δικά τους στα δικά τους μάντρα, χωρίς να βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα των γυναικών που προσπαθούν να συνδυάσουν τον ιδιωτικό με τον επαγγελματικό βίο. Και εδώ, στο Κοινοβούλιο. Να ξέρετε ότι είναι επιλογή των γυναικών. Θέλουν να κάνουν οικογένειες, θέλουν να κάνουν παιδιά και θέλουν να είναι και επαγγελματίε. Το να μην τις ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους, αυτό είναι καταπίεση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας αθαρρύνω να προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε λύσεις που πραγματικά να στηρίζουν τις γυναίκες. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, σας διαβεβαιώ κύριε, ακόμα και αν κυρωθεί, δεν θα λύσει τα προβλήματα των γυναικών, ούτε και αυτών που δουλεύουν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, τώρα συζήτηση. Ο κύριος Φαριά είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πορτογαλικά, αφού μπορώ να μιλήσω τη γνώσα μου, θα το κάνω. Τη μητρική και την πατρική μου γλώσσα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στον κύριο Πιμέντα Λόπες για το έργο του. Και συνδέεται και με αυτά που είπα και εγώ πριν. Ε. Πρόκειται για μια συνέχεια. Είναι δύο κείμενα τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή στο κείμενο και κυρίως στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία, να επεκταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι πολύ λεπτά ζητήματα, όπως λέω και εγώ στη δικιά μου την έκθεση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ε, διάφορες ευαισθησίες. Εγώ συμμετέχω σε μια πολιτική ομάδα για την οποία αυτά τα θέματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το κείμενο θα πρέπει να είναι συνενετικό, το κείμενο στο οποίο θα καταλήξουμε, για να μπορεί να στηριχτεί από όλες τις πολιτικές ομάδες τελικά. Επίσης, η συνάδελφος από το ECR που μίλησε πριν, υιοθέτησε μια συγκεκριμένη θέση. Και όσον αφορά τη δικιά μου τη χώρα, την Πορτογαλία, δεν θα σας πω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν γίνονται καλά και πολλά που γίνονται καλά όμως. Δεν έχουμε φτάσει στην τελειότητα, ίσως κάποια μέρα να την πετύχουμε την τελειότητα. Ελπίζω, τι να πω, ίνσαλα. Αλλά ίνσαλα στα το λέμε εμείς όχαλα. Μακάρι. Μακάρι λοιπόν να το καταφέρουμε. Οι αλλαγές αυτές να υλοποιηθούν. Αυτό θέλουμε. Μιλάω λοιπόν από το ΕΛΚ και έχουμε έναν συντάκτη γνωμοδότηση εδώ που είναι από την ΚΟΕ. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ μακριά από τον άλλον. Εκεί όμως πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε σύγκληση. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης όντως πρέπει ε, να κυρωθεί και όχι μόνο να τεθεί σε εφαρμογή. Και λίγες ε, χώρε που εντάξει δεν θα τι κατονομάσω τώρα αλλά που δεν έχουν κυρώσει ακόμα τη σύμβαση αυτή καλά θα κάνουν να το κάνουν, να βοηθήσουν οι συνάδελφοι, των οποίων οι χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή, να πιέσουν ώστε να γίνει. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και άλλα μέσα οργανώσει, εμπορικές συμφωνίες, συμφωνίες με τρίτες χώρες και ενισχύσεις που δίνονται σε άλλες χώρες πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και θα τελειώσω με το εξής. Θα ήθελα και για να παλαιώνουμε λίγο την ατμόσφαιρα μετά από τις επικρίσεις που ακούστηκαν, να γίνεται μνήα στα προβλήματα της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων και πιο συγκεκριμένα ε, σχετικά με τις ε, πιο καταπιεσμένες κοινότητες. Μετανάστες, καταπιεσμένη η ορολογία της αριστεράς. Το ξέρω, αλλά αυτή θα χρησιμοποιήσω. Και το φαινόμενο αυτό υπάρχει και στην Αμερική και στην Ασία. Θα ήταν καλό να προσθεθεί στο κείμενο. Τέλος, υπάρχουν καταστάσεις ακόμα και σκλαβιάς, πορνείας, καταναγκαστικής. Δυστυχώς όταν πήγα στην Κολομβία με την προσωπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είδα την κατάσταση στα σύνορα ανάμεσα στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα. Αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία με καταστάσεις σκλαβιάς. και καταναγκαστικής πορνείας. Είναι πραγματικότητα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν κάπως να συμπεριληφθεί και αυτό στο κείμενο. Παιδιά και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαρία. Η Άννα Μαρία Κορατσαμπίλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο συνάδελφος και να προσθέσω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ασχολείται με ένα ιδιαίτερα επικαιρό θέμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διότι βλέπουμε ότι η ακροδεξιά πηγαίνει χέρι με χέρι με πισωγύρισμα στα δικαιώματα των ε, γυναικών. Η ακροδεξιά, η σκληρή δεξιά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο επηρεάζουν την κυβέρνηση, τα δικαιώματα ε, και των γυναικών κινδυνεύουν, ε, συρρυκνώνονται οι οργανώσεις των πολιτών και από την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται μια γυναίκα να ανήκει στην ακροδεξιά χωρίς να σκέφτεται τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα της γυναίκας. Και να πω στην ε, συνάδελφο κυρία Βυσνιέσκα ότι γίνονται τα σεβαστές οι απόψεις της, διότι και αυτή η Ευρωβουλευτής είναι, έχει κάθε δικαίωμα να τοποθετηθεί ε, πάνω σε ένα σχέδιο έκθεσης. Δεν βλέπω βέβαια το πώς ε, συρρυκνώνονται τα δικαιώματά σας, ε, αυτό δηλαδή που είπατε, όταν ε, αναφέρεστε σε μια εκθέση την οποία δεν έχετε συντάξει εσείς. Σας παρακαλώ να μην είστε παράλογοι. Και να σας ρωτήσω κιόλα, έχετε πάει σε ένα κέντρο κακοποιημένων γυναικών, έχετε μιλήσει με γυναίκα που έχει βιαστεί, με ένα κορίτσι που είναι 13 χρονών, παντρεύτηκε καταναγκαστικά και είναι έγκυος, έχετε μιλήσει με μια γυναίκα που έχει ε, υποστεί ακροτηριασμό των ε, γεννητικών οργάνων. Αυτό σημαίνουν ε, δικαιώματα των γυναικών. Δεν έχει καμία σχέση με χριστιανικές αξίες, με το ότι είμαι περήφανη, που είμαι καθολική, οτιδήποτε. Έχει να κάνει με βία και η βία δεν είναι τίποτα άλλο από βία. Δυστυχώ, αυτές οι δυνάμεις που κινητοποιούνται ε, εκ των ε, έξω, ε, κινητοποιούνται και υποκινούνται μάλλον από άτομα σαν τον Πούτιν που οδηγούν σε Όπω είπα, συρρήκνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σου λέει, έσπασε στο πόδι σου, εντάξει τώρα, τι θέλει να πα στο νοσοκομείο. Ε, κινδυνεύουν από άτομα σαν τον Τραμπ, ο οποίο προσπαθεί να φημώσει τις ε, γυναίκες ε, στερούντας, ε, στερώντας τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα. Αυτό έχει καταφέρει κιόλα ε, ο Τραμπ με αυτό το φήμοτρο που έχει επιβάλει στις ε, γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και εκτός με τον Global Gag Rule. Βλέπουμε και στην Ευρώπη τι γίνεται όταν οι ακραίες πολιτικές δυνάμεις επιτίθενται στα, στην ισότητα και κυρίως στα δικαιώματα των γυναικών. Και γι' αυτό, για αυτούς όλους τους λόγους είναι τόσο σημαντική αυτή η έκθεση. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση, ότι υπάρχουν ακόμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπογράφουν τη Σύμφαση Κωνσταντινούπολης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με παρερμηνία και ως συνεισηγήτρια της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης δεν έχω σταματήσει να το λέω τα τελευταία ε, πέντε χρόνια. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν σαφέστατο ε, ως προς το τι σημαίνει έμφυλη βία. Είναι βία εναντίον των γυναικών ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο κρυμμένο, ούτε χριστιανικές αξίε ούτε δικαιώματα λότκι, ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με βία. Αλλά δυστυχώς ε, πολλοί αρνούνται να το ε, δουν αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να κινητοποιηθούμε. Ω προ το ψήφισμα τώρα, χρειάζεται να στείλουμε ένα έντονο μήνυμα στις γυναίκες και στις οργανώσεις των γυναικών ότι έχουν την πλήρη στήριξή μας, έτσι ώστε να αντισταθούν και να ε, προσπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Και μην ξεχνάτε ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Μην χρησιμοποιείτε ε, τα δικαιώματα των γυναικών για τους δικούς σας ιδεολογικούς ε, σκοπούς, για λιτότητα, επικουρικότητα κτλ. Μην χάνετε το μήνυμα το μήνυμα έχει να κάνει με τα δικαιώματα των γυναικών, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Η Τζούλι Ward θα πάρει το λόγο τώρα. Και σας παρακαλώ μέσα σε δύο λεπτά. Πολύ ωραία, όχι, θα είμαι σύντομη. Να επισημάνω ότι αυτό το πισωγύρισμα εμφανίστηκε το 1805 όταν δεν υπήρχε καν φεμινισμός γιατί το 1805 η καταπίεση εναντίον των γυναικών ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αυτή η λέξη λοιπόν backlash στα αγγλικά σημαίνει γυρίζω πίσω, πίσω γύρισμα και ποτέ δεν πρέπει να κοιτάζουμε προς τα πίσω αλλά πάντα προς τα εμπρός. Πρέπει αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, να παλέψουμε για να μην πάμε προς τα πίσω. Ας κατανοήσουμε λοιπόν την έννοια του πίσω γυρίσματος και ας μην φύγουμε από τον 21ο αιώνα για να γυρίσουμε προς τα πίσω. Επίσης, αυτό το πισωγύρισμα πολλές φορές ε, έχει αποτελέσματα ε, εξέγερσης. Έχετε δει τι έγινε στην Πολωνία με τις γυναίκες που βγήκαν στους δρόμους επειδή δεν ήθελαν να τους αφαιρέσουν τα δικαιώματά τους, να γίνει η ζωή τους δύσκολη, να κινδυνεύσει η υγεία τους. Αυτό συμβαίνει όταν προσπαθείς να γυρίσεις προς τα πίσω. Έχεις ε, τη συνέπεια ε, άνθρωποι που ποτέ μέχρι τότε δεν είχαν ε, πολιτικοποιηθεί να εξεγείρονται. Και ο Τραμπ κατά μία έννοια μας έκανε να ξυπνήσουμε και να αποκτήσουμε επίγνωση των κινδύνων γύρω μας, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, να πολεμήσουμε γι' αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε. Όταν δεν δημιουργούμε νομικά δεσμευτικά μέσα για να σταματήσουμε την έμφυλη βία, να σταματήσουμε τις απερβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο, ο κόσμος χάνει τη ζωή του. Πεθαίνουν γυναίκες, πεθαίνουν άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας συγχαίρω για την ε, ομιλία που μόλις κάνατε, για αυτά που μόλις είπατε, γιατί ξέρετε και εγώ συναντήθηκα με αυτές τις γυναίκες οι οποίες ήταν αποδέκτες βίας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπήκα στην πολιτική. Βρίσκομαι εδώ ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς εξαιτίας της οδύνης που βίωσαν αυτές οι γυναίκες και οι οικογένειές τους. Και νομίζω πως ε, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες όλοι μαζί, να αγωνιστούμε ε, και να δούμε ότι εάν δεν δεσμευτούν τα κράτη-μέλη, όχι μόνο υπογράφοντα τη δήλωση, αλλά και ε, κυρώνοντά τη και επενδύοντα σε αυτήν, παρακολουθώντα την εφαρμογή τη, ε, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να τα κάνουμε όλα. Είναι ολόκληρη η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ, Βυσνεύσκα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι εξοργισμένη Γιατί ακούστηκε ότι είμαι υπέρ της βίας κατά των γυναικών. Δεν ξέρω αν αυτή αυτό που άκουσα ως μετάφραση. Λοιπόν, θα ξαναπώ αργά και καθαρά. Είμαι κατά της βίας. Είμαι κατά της βίας. Τώρα λέει κανείς ότι αυτή είναι η θέση της δεξιάς. Τον αποδίδει κανείς τέτοιε κατηγορίες, ανθρώπους που απλώ είναι κατά των αμβλώσεων και κατά τη ευθανασία, αποτελεί παραλογισμό. Είμαι κατά της βίας. Και παρακαλώ να μην μου αποδίδετε τέτοιες ιδέες. Για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, έχω από το εξής. Εάν το φύλλο ορίζεται και κοινωνικά και, φιλετικά. Ε, διαφωνώ, διαφωνώ. Αν βάλουμε και άλλους παράγοντες, δηλαδή με πολιτιστικούς μάλλον κλπ. Αυτά είναι αριστερή φιλολογία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι από την Πολωνία. Η βία κατά των γυναικών στην Πολωνία είναι από τις χαμηλότερε στην Ευρώπη. Δείτε το αν θέλετε. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Όχι, δεν θα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά από την αρχή, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ένα λεπτό για τον εισηγητή, παρακαλώ. Πολύ γρήγορα, κυρία Πρόεδρε. Η σύντομη σημερινή συζήτηση είναι προανάκρους με αυτόν που θα ακούσουμε και θα πούμε τις επόμενες μέρες. Ας πάρουμε στα χέρια μας πρώτα το τελικό κείμενο του ψηφίσματος. Κοιτάξτε, εγώ δεν ε, διαφωνώ ότι υπάρχει επιστοδρόμηση, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που έχουν κάνει διάφορες κυβερνήσεις. Κάποιες τέτοιε επιλογές, αποφάσεις είναι οικονομικές. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ξέρετε, η ακροδεξιά. Εγώ απορρίπτω αυτή την άποψη ότι φταίει μόνο η ακροδεξιά και γι' αυτό παρατηρούμε οπισθοδρόμεις. Και όμως, κεντρώες κυβερνήσεις, προοδευτικές κυβερνήσεις έχουν συμβάλει και αυτές στην υποχώρηση, στην οπισθοδρόμηση. Ας πούμε, μέσω οικονομικής πολιτικής, στην οπισθοδρόμηση των οικονομικών δικαιωμάτων. Για να μην μιλήσουμε για τη μετανάστευση γυναικών από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο και ο συνάδελφος Φαρία προηγουμένως. Και ακούστε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Ένα σχολείο για την πορνεία. Και βέβαια είπε κάποιο εξαναγκασμένη ε, υποχρεωτική, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει εξαναγκασμένη ή μη πορνεία. Ε, και αυτό βέβαια μια άλλη κουβέντα. Το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινή βάση, να συμφωνήσουμε μεταξύ μας, ώστε το ψήφισμα να, γίνει, να εγκριθεί με την ευρύτερη δυνατή συνένεση από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Αντί να αναλωνόμεθα για μια φορά σε στρατηγικές και νόμους κλπ. Λοιπόν, τώρα για την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το θέμα είναι όλα αυτά να υλοποιούνται στην πράξη. Πρόεδρος. Λοιπόν, προθεσμία ε, τροπολογιών. 4 ε, Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι. 4 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι. Έχετε μερικέ μέρε μπροστά σα η υποβολή τροπολογιών. Η ψηφορία στην Επιτροπή μα είναι 8 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια πάμε 2 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ όλου του ε, σημαντικούς συμμετέχοντες. Α, επόμενη συνάντηση. 10 Οκτωβρίου. Επόμενη συνεδρίασή μας. Ξεκινάμε 8.30. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς που έμειναν λίγα λεπτά μαζί μας. Γεια σας.